Το σχέδιο ημερήσια διάταξη εστάλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 12 Μαΐου. Θα πρέπει να έχετε αντίγραφο στους φακέλους σας. Έχουμε έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 22-23 Μαρτίου. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Έχουμε την, ε, έχουμε διερμηνία στις ε, συνήθεις Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι μία παρουσίαση του Επιτρόπου Σεμέτα, ο οποίος ε, θα μιλήσει για τον, ε, οποίος θα μιλήσει για, την, ε, για τον πρώτο μήνα των δραστηριοτήτων του στον τομέα της φορολογίας της Ελληνικής Ένωσης του έλεγχου και της καταπολέμησης της απάτης. Θα ήθελα να του δείσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Χαίρομαι που μπορώ σήμερα να σας ε, παρουσιάσω σήμερα ε, το πρόγραμμά μου για την φορολογία, την Τελωνική Ένωση, τον έλεγχο και την ε, καταπολέμηση της απάτης. Έχω ετοιμάσει την ατζέντα αυτή σε συνεργασία με την Επιτροπή σας για να πετύχω τον στόχο, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει να ε, εμποδίσουμε τα λάθη από την ε, κακή δημοσιονομική διαχείριση και την καταπολέμηση οποιοδήποτε είδους απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους ε, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την ε, απαλλαγή και τον ε, λογιστικό έλεγχο, θα ήθελα να ε, πω ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά μέσα σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο. Ο κίνδυνος λαθών αυξάνεται με την πολυπλοκότητα των κανόνων. Γι' αυτό, ακολουθώντα τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και τα ψηφίσματα της ε, αρχής για την απαλλαγή, η Κομισιόν ε, ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, την απλοποίηση για τις παροχές και τους κανόνες για την επιστροφή. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολη η, ε, ε, οικονομική διαχείριση, ε, διατηρώντας όμως τις αρχές για την οικονομική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετηθεί πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα για τα αποδεκτά περιθώρια λάθους σε διάφορους τομείς. Ε, αυτό θα σπληρωθεί ε, από τους υπόλοιπους ε, τομείς πολιτικής μέχρι το 2011. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση που βασίζεται στις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου θα σημάνουν πιο αποτελεσματική πολιτική ελέγχου στα διάφορα προγράμματα. Παράλληλα θα προωθήσω ποιοτική προσέγγιση όσον αφορά τις δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η και ε, η ε, κανονικότητα στις συναλλαγές ε, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Μου φαίνεται όμως σημαντικό να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Θα επικεντρωθούμε στην απόδοση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συμπεριλάβουμε σαφείς στόχους και δείκτες ε, κατά την εκπόνηση των ε, νέων προγραμμάτων δαπανών. Επίσης, θέλω να ενισχύσω το ρόλο της ε, του εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, όπως φαίνεται και από τις συστάσεις για την χορήγηση απαλλαγή έχω ζητήσει από την Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου να αναπτύξει μεθοδολογία όχι μόνο για να ελέγξει αν οι στόχοι ε, που αναφέρονται στις συστάσεις εφαρμόζονται, αλλά και αν τα μέτρα που αναλαμβάνονται ε, μετριάζουν τον κίνδυνο. Τέλος, πρότεινα να συμπεριλάβουμε στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού μία ε, διάταξη για τα ευρωπαϊκά trust funds ώστε να διασφαλίζουμε την πολυμερή ε, συνεισφορά ε, σε περιπτώσεις ε, όπως για παράδειγμα των εξωτερικών δράσεων. Αυτό όχι μόνο βελτιώνει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ενισχύει και το ρόλο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Χρειαζόμαστε μια νέα εταιρική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι καταλαβαίνουν το ρόλο τους και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για να πετύχουμε τους κοινούς μα στόχους. Αυτό μεταφράζεται ιδιαίτερα με απαιτήσει για αιτήσια δήλωση διασφάλισης από του, τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών. Η δήλωση αυτή θα αποτελεί αντικείμενο εξέταση σε του Συμβουλίου Ελέγχου. Παράλληλα θα εξετάζουμε την προστιθέμενη αξία των ε, εθνικών περιλήψεων ε, όσον αφορά την, την διασφάλιση από πλευράς της Επιτροπής. Οι εθνικές αρχές ε, ελέγχου θα ε, κληθούν να συμμετέχουν περισσότερο στον, ε, στην εφαρμογή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Όπως προτάθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2004. Τέλος, θα συνεργαστώ ε, για την ε, οργάνωση διάσκεψης για όλους τους ενδιαφερομένους που ε, έχουν να κάνουν με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαδικασίας του, της απαλλαγής όπως φαίνεται από το ψήφισμα του 2008 για την απαλλαγή. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2011 για να μπορούμε για να μπορεί η Επιτροπή να αναλάβει την ε, δημοσιονομική της ευθύνη κατά την εκτέλεση του ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη πληρωμή θα πρέπει να υπάρχουν επαρκεί και εξαντλητικέ πληροφορίε, όχι μόνο όσον αφορά του τομεί για του οποίου είναι άμεσα αρμόδια η Επιτροπή, όπω είναι η άμεση διαχείριση, αλλά και όσον αφορά το τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό οι πληροφορίες για την ανάκτηση και τις ε, δημοσιονομικές κινήσεις ε, στους ε, λογαριασμού θα βελτιωθούν. Για τα γεωργικά και διαφορετικά ταμεία θα υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία ανά κράτο μέλο. Θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση των κρατών μελών όσον αφορά τι δημοσιονομικέ διορθώσει, όπου έλεγχη, συστάσεις, κατάρτιση και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση αν θέλουμε το, ελεγκτικό συνέδριο να λάβει υπόψη την ε, πολιετή διάσταση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ε, στραφώ στο άλλο μέρος ε, του χαρτοφυλακίου μου, την ε, καταπολέμηση της απάτησης και τον Όλαφ. Η πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης και ο Όλαφ παίζουν σημαντικό ρόλο σε εποχές οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό οι πόροι να δαπανώνται με το σωστό τρόπο. Η απάτη και η διαφθορά θα πρέπει να εντοπίζονται και να αποτρέπονται. Θα πρέπει επίσης ε, να ανακτώνται οι χαμένοι πόροι. Γι' αυτό ο Όλαφ ε, χρειάζεται ε, αυξημένη προσοχή από την πλευρά μου, την οποία και θα έχει. Τα επόμενα θέματα του προγράμματός μου θα τα έχετε ήδη λάβει γραπτός, αλλά θα ήθελα να σας τονίσω τα εξής. Όσον αφορά τον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ, είναι σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα για να βρούμε νέο Γενικό Διευθυντή προτεραιότητα είναι να βρούμε τον καλύτερο υποψήφιο για τη θέση αυτή. Θα σας στείλω σύντομα το ε, προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αυτή και προσλέπω στην ε, ενεργό συμμετοχή σας στη διαδικασία αυτή. Όσον αφορά τον ορισμό της Εποπτικής Επιτροπής του Όλαφ ε, στις 25 Μαΐου έστειλε επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό όπως ε, συμφώνησαν, καθότι συμφώνησαν όλα τα μέλη ε, να ε, συμμετάσχουν σε δεύτερη θητεία, προβλέπεται ο διορισμός του. Η θητεία του σε λίγη στις 30 Νοεμβρίου του 2011. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί σας και με το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Η διαδικασία επιλογής για μια νέα εποπτική ε, αρχή θα πρέπει να ε, ξεκινήσει εγκαίρως. Τρίτον, αναθεώρηση του Όλαφ. Όπως ε, είπα και στην ακρόασή μου, είναι προτεραιότητα να προωθήσουμε το έγγραφο για την αναθεώρηση του Όλαφ. Ε, θα παρουσιαστεί σε εσά και στο Συμβούλιο πριν τις θερινές διακοπές. Ε, με βάση ε, διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πάνω στο έγγραφο αυτό, η Κομισιόν θα παρουσιάσει αναθεωρημένη πρόταση. Ειλικρινά ελπίζω ότι με τη βάση αυτή η νομοθετική διαδικασία της αναθεώρησης του Όλαφ θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Τέταρτον, βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Όλαφ. Πέρα από την αναθεώρηση της νομικής βάσης του Όλαφ, η Κομισιόν θα επιδιώξει περαιτέρω βελτίωση ε, της αποτελεσματικότητας ε, του Όλαφ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ε, συστάσεις της Εποπτικής Επιτροπής, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη συνέχεια της σε ελέγχου της του 2005. Θα συναντηθώ και με την Εποπτική Επιτροπή. Επίσης θα εξετάσω περαιτέρω τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε διοικητικό επίπεδο και στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού του Όλαφ. Πέμπτον, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την προετοιμασία της ε, δημιουργίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για την προστασία του των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το θέμα αυτό απαιτεί εις βάθος συζήτηση για να, ε, για να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον Όλαφ. Η Αντιπρόεδρος Ρέντιν και εγώ ζητήσαμε τις ε, υπηρεσίες σας να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει ε, στη ε, διαδικασία αυτή και η Κομισιόν βασίζεται στην συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή ε, πρωτοβουλία που θα βελτιώσει σε βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιβολή του νόμου. Ε, επίσης, ε, θα φροντίσω να ε, εφαρμόζονται τα διεθνή μέσα και να αναπτυχθούν περαιτέρω για να καταπολεμήσουμε για παράδειγμα το λαθρεμπόριο σιγάρων και άλλα τέτοια πράγματα και άλλα τέτοια θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται ένα λειτουργικό πλαίσιο. Ανέφερα ως ε, παραδείγματα, κάποιες ε, διατάξεις ε, που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες συμφωνίες συνεργασίας, εταιρικής σχέσης. Έχουμε διάσκεψη στον Παναμά τον Οκτώβριο του 2010 και η οποία ε, έχει ως αντικείμενο Διεθνή Συμφωνία για την ε, καταπολέμηση του ελευθερμπορίου των ε, τσιγάρων. Επίσης το θέμα της φοροδιαφυγής είναι πολύ σημαντικό. Θα μιλήσω με τους Προέδρους του Συμβουλίου για να φροντίσω να παραμείνει το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό είναι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Λίχτενστάιν όσο γίνεται πιο γρήγορα για την καταπολέμηση της απάτης. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην γενική πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης η συνεργασία ανάμεσα στον Όλαφ και κάποιες γενικές διευθύνσεις θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός της ε, Επιτροπής. Κάποιες υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη στρατηγική αντικαταπολέμηση της απάτης, όχι όλες όμως. Ο Όλαφ ε, έχει αρχίσει να ετοιμάζει αξιολογήσεις ε, κινδύνου για διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, αλλά αυτά είναι μόλις η αρχή. Γι' αυτό Χρειάζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για στρατηγικές καταπολέμησης απάτης εντός της Κομισιόν. Ε, αυτές θα αναπτυχθούν ε, κατά τη διάρκεια της θητείας μου που να αφήνουν χώρο για ε, διάφορα μέσα που να είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και θα πρέπει να παρουσιαστεί σε νέα ανακοίνωση της επιτροπή. Θα ε, σας ενημερώνω τακτικά για τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Ε, βασίζομαι στην υποστήριξή σας για να εφαρμόσουμε την ημερήσια αυτή διάταξη ε, στο πνεύμα της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για, την, για τις πραγματικά εντυπωσιακές εξαγγελίες και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά τροποτινά παρουσιάζεται ένα πενταετές ε, πρόγραμμα. Αυτό κάνει μια πολύ καλή εντύπωση θα έλεγα. Αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να σε επισημάνω ότι δεν πρόκειται παρά για εξαγγελίες και μπορούμε να αποτολμήσουμε ε, ε, να πούμε ότι περιμένουμε, ότι γνώμονας για τις εξεγγελίες αυτές θα είναι οι πραγματικές δράσεις, τουλάχιστον ο γνώμονας της δικής μας πολιτικής ομάδας του ΕΛΚΑ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε στο τέλος, γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένο. Είπατε ότι εντός της Κομισιόν η καταπολέμηση της απάτης και η πρόληψη θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρότερα τώρα υπόψη από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και η καταπολέμηση της απάτης στην Κομισιόν θα πρέπει να προσλάβει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχε μέχρι τώρα και αν ε, ε, ε, μας παρουσιάσετε το έγγραφο εργασίας στην αναθόρυση της Όλαφ. ελπίζουμε σε αυτό να συμπεριλαμβάνονται και δικές μας προτάσεις όταν μας το παρουσιάσετε. Κατά τα άλλα, όπως σας είπαμε, είπατε πολλά. Ε, και αν δούμε τι γίνεται στην πράξη όσον αφορά τη βελτίωση της δήλωσης αξιοπιστίας ειδικότερα, θα πρέπει να το συνδυάσουμε με τις νέες ρυθμίσεις, ούτως ώστε κάποια πράγματα να λύνονται αυτόματα με τη βοήθεια των νέων κανόνων. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία μετρούσαν μέχρι τώρα δεν μετρούν ε, πια. Υπάρχουν λοιπόν, εψέρχονται λοιπόν αυτόματα κάποιες βελτιώσεις βάσει του νέου δικαίου και όχι χάρη κάποιων επιπρόσθετων δραστηριοτήτων. Για μα, δύο πράγματα είναι σημαντικά. Τι θα γίνει στη συνέχεια με την Όλαφ. Είπατε ότι θέλετε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα τη Όλαφ και θα έχει πραγματικά ένα νόημα να μα πείτε πώ θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί η Όλαφ έχει πολλά προβλήματα, οι χρονοβόρες διαδικασίες, το σύνθετο νομικό περιβάλλον, οι εξαιρετικά απρόθυμες χώρες μέλη, όταν το ζητούμενο είναι τα αποτελέσματα τη Όλαφ να εφαρμοστούν νομικά. Και θα ήθελα να σα επισημάνω ότι τα ελλειπή στατιστικά στοιχεία, γιατί μόνο 7% των περιπτώσεων οδηγούν σε πραγματικές καταδίκες, τελικά θα πρέπει να υπαχθούν σε κάποιον έλεγχο. Γιατί νομίζω ότι δεν θα βελτιωθεί με τον τρόπο αυτό η αποτελεσματικότητα. Τι προτείνετε να κάνετε, πώς θέλετε να επηρεάσετε τις χώρες μέλη ή το ανεκτό περιθώριο σφάλματος ο... Ε, ε, μου διαβάσετε αυτά τα έγγραφα μαζί με τον κύριο Λεβαντόσκι όσον αφορά τις εκτελεστικές ε, διατάξεις. Και αν δούμε τι γίνεται με αυτό τον ανεκτό κίνδυνο, το περιθώριο αποδεκτού σφάλματος, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι σωστό ότι μας πετάτε το μπαλάκι. Λέγοντας το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί σχετικά. Εγώ αισθάνομαι κάποια μηχανία και θα πρέπει να πω ότι δεν τα φαντάστηκα μέχρι στιγμής έτσι τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να γίνει θα πρέπει να προηγουμένως να οριστεί ακριβέστερα, να γίνει πιο συγκεκριμένο. Η έκθεσή μου είναι ολοκληρωμένη και δεν έχει γίνει τίποτα. Ενώ είναι σημαντικό εδώ να γίνουν κάποια βήματα προς τα μπρος. Γιατί κάθε μέρα που χάνομαι είναι υπέρ των όσων φοροδιαφεύγουν. Και νομίζω ότι τίποτα δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Γιατί το Συμβούλιο τελικά δεν αποδέχεται ούτε καν αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι. Νομίζω λοιπόν ότι θα είχε νόημα η Κομισιόν να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση και να συμπεριλάβει και εμάς, γιατί εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, κύριε Επίτροπε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στου στους πολίτες. Και δεν μπορώ παρά να σα ενθαρρύνω πραγματικά να κινηθείτε προ αυτόν τον δρόμο, αλλά πραγματικά να το κάνετε ε, με την απαιτούμενη ενέργεια και όντα πιο συγκεκριμένος. Γιατί αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ ισχνά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, το ελεκτικό συνέδριο με τις εκθέσεις του μας δείχνει ότι η εποπτεία όσον αφορά τα ταμεία της Ένωσης δεν είναι πάντα ούτε αποτελεσματική ούτε πολύ καλή. Γι' αυτό και τα ταμεία δεν χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο επικροτώ την πρότασή σας για εθνικές δηλώσεις. Χρήσιμη θα είναι στο μέλλον για διάφορα προγράμματα και την αποδοτική χρήση τους στα κράτη-μέλη. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα για την ανάκτηση κονδυλίων στην περίπτωση λαθών ή κατάχρησης. Και το ερώτημα είναι Πώς θα βελτιώσετε την υποπτία των προγραμμάτων. Θα ήθελα συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο να απαντήσετε στα... στους δύο βουλευτές. Thank ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ευχαριστώ την κυρία Γκρέσλε που υποστηρίζει την ημερήσια διάταξη που σας παρουσίασα. Μιλάμε για εφαρμογή. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι εμείς αυτό που υποσχεθήκαμε το κάνουμε. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε δύο προτάσεις για το δημοσιονομικό κανονισμό. Ανακοίνωση της Κομισιόν για το ανεκτό περιθώριο λάθους. Είχαμε πει το Μάιο, έγινε το Μάιο. Για την έννοια αυτού του ανεκτού περιθωρίου λάθους, ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει το νομικό πλαίσιο της έννοιας αυτής. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα έρθει μετά από τη συζητήση που θα γίνει για τις ε, προτάσεις με βάση την ανακοίνωση. Εκεί υπάρχει μια λεπτομερής ανάλυση της έννοιας αυτής κατά τομέα. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επομένως θα πάρουν πλήρες μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και τα δύο σκέλη της αρχής του προπολογισμού με τις συζητήσεις θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για το ανεκτό περιθώριο λάθους στους ε, τομείς που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Όλαφ. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Έχουμε το έγγραφο μελέτης ή περισυλλογής, στο πούμε reflection paper. Το κείμενο, το έγγραφο αυτό ακριβώς αναφέρεται στα θέματα που εσείς θίξατε. Νομική βεβαιότητα, συμμετοχή των κρατών μελών. Τώρα το, η χρονική διάρκεια των διαδικασιών αποκινούμε την Όλαφ και με το ελεκτικό συνέδριο το οποίο αναλύει την κατάσταση και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ να βραχυνθούν οι διαδικασίες αυτές χρονικά όσον αφορά την Όλαφ γιατί πραγματικά καθυστερούν σε πολλές περιπτώσεις. Χρειάζονται σαφείς κανόνες. Να βραχυνθεί η χρονική τους διάρκεια. Και πρέπει να γίνονται τακτικά αναφορές κατά περίπτωση όταν σημειώνεται η υπέρβαση του χρονικού ορίου που έχει δοθεί. Επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή της εποπτικής αρχής. για να γίνει η κατάσταση όσον αφορά τις διαδικασίες και τη διάρκεια των διαδικασιών πιο αποτελεσματική. Συμφωνία με τον Λίχτενστάιν. Ξέρετε ότι αυτό είναι τμήμα του πακέτου που συζητάμε στο Συμβούλιο. Είναι μερικές οδηγίες για συνεργασία σε θέματα φορολογίας η περίφημη οδηγία για τη ε, αποταμίευση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών Όντως η πρόταση έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο από δύο κράτη-μέλη Αύριο θα πάω στη Γερμανία για να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Υπουργό Σόιμπλε και ελπίζω να βρεθεί η λύση. Πρέπει οι συμφωνίες αυτές και όλο το πακέτο και την χρηστή διακυβέρνηση πρέπει να εγκριθεί σε επίπεδο ένωσης. Διότι μόνο μετά θα μπορούμε να προωθήσουμε την χρηστή διακυβέρνηση διεθνώς. Βέβαια, τα κράτη-μέλη χρειάζονται πόρους για την καταπολέμηση της φοραπάτης και φοροδιαφυγής. Ανάκτηση κονδυλιών. Υπάρχουν δύο είδη. Η ανάκτηση σε επίπεδο ένωσης Ήδη με τις ε, οικονομικές εκθέσεις του 2009 θα έχετε πληροφορίες για αυτού του είδους την ανάκτηση κατά κράτος μέλος και θα μπορείτε να κάνετε και σύγκριση. Η δε ανάκτηση σε επίπεδο κράτους μέλους οριστικοποιούμε τους ε, επιτόπιους ελέγχους, spot checks στα κράτη-μέλη, να δούμε πώς δουλεύει το σύστημα. Όλα τα κράτη-μέλη θα τα κοιτάξουμε και με βάση τους ελέγχους αυτούς θα κάνουμε συστάσεις. και ανταλλαγή της, των άριστων μεθόδων μεταξύ των χωρών. Αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γερμπράντι. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίαση του εγγράφου το οποίο μας εστάλει εκ των προτέρων. Βρίσκω ότι είναι πολύ καλή αρχή αυτή και ελπίζω ότι έτσι θα βελτιωθούν πολλά πράγματα. Κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν το θέμα είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και αργότερα θα λάβουμε και σχετική ανακοίνωση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να τη δούμε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη-μέλη διαθέτουν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ε, εδώ θα ήθελα να κάνω μια επίκριση. Βρίσκω ότι είσαστε πολύ προσεκτικός, επιφυλακτικός εδώ. Πιστεύω ότι θα μπορούσατε να επιδείξετε περισσότερη συνέπεια. Είσαστε αρκετά προσεκτικό στον τομέα αυτών και θέλετε να στηριχτείτε στις εμπειρίες των κρατών μελών. Βλέπουμε όμως ότι τα κράτη-μέλη ε, βλέπουν όλο και πιο επικριτικά τις δημόσιες δαπάνες και αναρωτιέμαι μήπως ήρθε η ώρα να εξετάσουμε επικριτικά και τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μην ξεχνάμε είναι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ευρώπης. Μήπως λοιπόν έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή να ενεργήσουμε εδώ πιο δραστικά και όχι τόσο προσεκτικά όσο προτείνετε εσείς. Και σκέφτομαι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο ε, το αν είναι σωστή η, ε, η πληρωμή των δαπανών αυτών, αλλά να εξετάσουμε και την αποτελεσματικότητα. Ο κύριος... Ο κύριος Γκάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ πλήρες το πρόγραμμα εργασίας σας ε, και εάν καταφέρετε να εφαρμόσετε όλα αυτά που λέτε θα έχουμε προχωρήσει στον τομέα της εφαρμογής του προϋπολογισμού ε, της Ευρώπης. Ε, ερώτηση για το σημείο 7, εξωτερικές δράσεις. Ε, Κάτα την απαλλαγή διαπιστώσαμε μεταξύ άλλων, διότι Ακούσαμε και στις ακροάσεις των επιτρόπων κατά την απαλλαγή ότι η υποβολή εκθέσεων από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ικανοποιητική όσον αφορά του σπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η έκθεση του συναδέρφου Μπόχουσλαβ ε, Λιμπεράτσκι ήταν και ιδιαίτερα επικριτική. Στο ε, σημείο 7 λοιπόν βλέπουμε κάποια σημαντικά μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνετε σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κύριο Σκυλακάκης. Uh, Επίτροπε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις πολιτικές που προτείνετε για τον Όλαφ και το γεγονός ότι θα επανεξετάσετε τρόπους ενίσχυσης του Όλαφ. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το ποσοστό των υποθέσεων που οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ε, υποθέσεων που ξεκινούν καθώς ε, και τον αριθμό των ε, ερευνητών του Όλαφ, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πολλές απάτες και έχουμε αδύναμο σύστημα καταπολέμησης της απάτης. Οι ερευνητές βρίσκονται στην καρδιά του συστήματος αυτού. Έχω κι εγώ μια ερώτηση. Σε σχέση με αυτό που μας λένε τα αρμόδια όργανα μεταξύ των οποίων και η Όλαφ, το ελεκτικό συνέδριο και εμείς το διαπιστώσαμε άμεσα εξάλλου τι είδους πολιτική θεσμική δραστηριότητα σκοπεύει να ασκήσει η Κομισιόν έναντι των κρατών μελών που όλο και πιο σταθερά παρατηρούνται παρανομίες και απάτες όσον αφορά τα δημόσια κονδύλια και όλο και πιο μεγάλη διαφθορά. Και μαφίες θα έλεγα που εποφελούνται από δις ευρώ που δίνονται σε ορισμένα κράτη μέλη. Τι πολιτική πρωτοβολία σκοπεύετε να πάρετε εσείς και η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω τα ερωτήματα τα οποία Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που συμφωνείτε με την βασική αρχή της απλούστευσης. Και θα έλεγα ότι στο δημοσιονομικό κανονισμό ε, προτείναμε να παραμείνουν 100 άρθρα από τα 800 που είναι αυτή τη στιγμή και πολλά που προτάθηκε να αλλάξουν θα οδηγήσουν σε σημαντικές απλουστεύσεις στο δημοσιονομικό κανονισμό. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι θέσαμε το ζήτημα αυτό στην το τομεακή νομοθεσία. Γι' αυτό προτείναμε και μία απλούστευση στο σχετικό δημοσιονομικό κανονισμό. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία, προτείνουμε στο δημοσιονομικό κανονισμό την εφαρμογή ετήσιων δηλώσεων διαχείρισης στο επίπεδο των ενδειγμένων οργάνων, τα οποία να τα ελέγχουν ανεξάρτητοι ελεγκτικοί οργανισμοί. Πρόκειται λοιπόν για ένα μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στη Γεωργία και το οποίο αποδείχθηκε ότι λειτουργεί σωστά και οδήγησε σε βελτιώσεις στον τομέα της γεωργίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. και αν ε, συμφωνήσετε, γιατί ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει βεβαίως ε, να εγκριθεί στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ε, συναπόφασης με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το μοντέλο αυτό των ετήσιων δηλώσεων διχείρισης θα βελτιώσει το επίπεδο λογοδοσίας των χωρών μελών όσον αφορά την χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Τώρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, το έχω ήδη αναφέρει στην ομιλία μου, είπα ότι συμμερίζομαι πλήρως τη δική σας άποψη ότι δεν αρκεί να ελέγχουμε την επιλεξιμότητα των δαπανών, κάτι το οποίο βεβαίως είναι επίσης σημαντικό σε σχέση ακριβώς με την ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Και αυτό θα το προσεγγίσουμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εξωτερικής ε, ελεγκτικής υπηρεσίας. Και ζήτησα από την υπηρεσία αυτή, την ελεγκτική αυτή υπηρεσία, όταν διενεργούν αυτούς τους ελέγχους, να μην το κάνουν σε σχέση με την χρησιμοποίηση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η χρήση των κονδυλίων και επίσης κατά πόσο χρησιμοποιούνται κάποιοι δείκτες αποδοτικότητας βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα ούτε ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να μελετήσει αυτούς τους ε, δείκτες αποδοτικότητας για να μελετήσει και την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης αυτών των κοινοτικών κονδυλίων. Τώρα, όσον αφορά τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, ένα σημαντικό στοιχείο είναι το ότι στο πλαίσιο του λογιστικού συστήματος της Επιτροπής δημιουργήσαμε κάποιους δείκτες που σχετίζονται με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και αυτό θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγης του τι ακριβώς κάνουν οι μη κυβερνητικέ οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν στην, στα κοινοτικά αυτά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί ο βαθμός διαφάνειας σε αυτό το τομέα. Και επίσης θα δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό trust fund. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και συμπεριλαμβάνεται ήδη η πρόταση αυτή στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και εφόσον εγκριθεί τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση όχι μόνο να παράσχει τη δική της ε, υποστήριξη μέσω των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα μπορέσει να οργανώσει και τη δική της υποστήριξη μέσω των δικών της Trust Funds. Και έτσι τα προβλήματα όσον αφορά τη μετάδοση πληροφοριών ή της πρόσβασης στις πληροφορίες θα επιληθούν. Γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε τους δικούς μας, να καθορίσουμε τους δικούς μας ε, ελέγχους σύμφωνα με τα δικά μας ε, συστήματα. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική υπηρεσία δράσης, την υπηρεσία εξωτερική δράση, συγγνώμη, είπα ότι οι επιχειρησιακέ δαπάνε ε, παραμένουν γράφονται στον προπολογισμό τη Επιτροπή και η απαλλαγή θα αφορά την υπηρεσία ε, και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα υπάρξει μια ξεχωριστή απαλλαγή, διαδικασία απαλλαγή, η οποία όμως επίση θα υποβληθεί σε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι το κοινό μας συμφέρον να παραμείνει υπόλογη η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης στην ε, αρχή, στην υπηρεσία απαλλαγή. Όσον αφορά τώρα την Όλαφ και τον αριθμό των ε, ανακριτικών διαδικασιών, θα έλεγα ότι κάποιοι αριθμοί που αναφέρονται συχνά, ότι μόνο, που ανέφερα και εγώ, ότι μόνο 7% όλων των περιπτώσεων οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ίσως δεν είναι απολύτως ακριβή αυτά τα στοιχεία. Και θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτή τη στιγμή. Έχουν ολοκληρωθεί οι ανακριτικές αυτές διαδικασίες. Η πραγματική αριθμή λοιπόν είναι υψηλότερη. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της Όλεφ. Ξέρετε ότι εγώ εργάζομαι μόνο εδώ και τρεις ε, μήνες, άρα δεν μπορείτε να περιμένετε ε, μέσα στο διάστημα αυτό να επιληθούν όλα τα προβλήματα με την Όλαφ. Αλλά στο πλαίσιο της αναθεώρησης ή στην ε, προπαρασκευή αυτού του εγγράφου προβληματισμού, του κειμένου προβληματισμού όσον αφορά τα προβλήματα αποτελεσματικότητας της Όλαφ, αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στα εργαλεία που θα επιτρέψουν μια αύξηση της αποτελεσματικότητας. Και ελπίζω οι προτάσεις αυτές να τύχουν της δικής σας υποστήριξης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε το δεδειγμένο νομικό πλαίσιο που θα που θα αυξήσει, μια, που θα αυξήσει το βαθμό αποτελεσματικότητας. Το ίδιο ισχύει και για το ετήσιο διαχειριστικό πρόγραμμα και πιο λεπτομεριακά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τα οποία επιβάλλονται στην ε, Κομισιόν. Ζήτησα από τις υπηρεσίε να καταρτήσουν, να ορίσουν μάλλον συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά τη διάρκεια των ανακρίσεων ή των ερευνών, την μορφή συνεργασίας με τις χώρες μέλη κλπ. Και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της δικής μου εντολής η αποτελεσματικότητα της όλα θα αυξηθεί σημαντικά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κοινό μας συμφέρον. Όσον αφορά τώρα την ε, απάτη, τις απάτες που έχουν εντοπιστεί, η απάντηση εδώ είναι αρκετά απλή. Η Επιτροπή εφαρμόζει μηδενική ανοχή έναντι της απάτης. Και αυτό που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσουμε να απαλλάξουμε την Όλαφ από ελάσσονα ζητήματα και να τα αναθέσουμε σε άλλα όργανα ούτω ώστε η Όλαφ να μπορέσει να επικεντρώσει τις δικές της δραστηριότητε σε πραγματικά ουσιαστικά θέματα σε θέματα βαρύνουσας σημασίας και σημαντικές περιπτώσεις. Αυτό θα επιτρέψει μια καλύτερη αξιοποίηση του ανακριτικού ερευνητικού δυναμικού. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους αύξησης της αποτελεσματικότητας της Γκρέσιλε. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Το γεγονός ότι η Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή δεν ε, ε, ασχολείται πολύ με τον όλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν παρατηρούμε προσεκτικά τι γίνεται εκεί. Κύριε Επίτροπε, και εσείς θα πρέπει σύντομα να μας παρουσιάσετε αποτελέσματα στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα της πίστης των κρατών μελών έχει ε, φανεί με την ε, οικονομική κρίση. Δεν θα πρέπει να ε, τρέχουμε αυταπάτες. Τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν πάντα πολύ πιστά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε συχνά διαμάχες με τα κράτη-μέλη και γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα να φύγετε από την αίθουσα ε, γνωρίζοντας ότι έχετε την ε, υποστήριξή μας, αλλά την υποστήριξή μας για να δούμε αποτελέσματα. Ε, όταν βλέπουμε τι έχει υποβληθεί εδώ, κάποια πράγματα πάντα ήταν σημαντικά για μας. Αυτό το γνωρίζει η Κομισιόν, για παράδειγμα το θέμα των εθνικών δηλώσεων. Και βλέπω στον δημοσιονομικό κανονισμό ότι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ε, εθνικές δηλώσεις μέχρι το 2015. Έχουμε περιλήψεις οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό προβληματικές. Οι περιλήψεις αυτές μέχρι τώρα είναι σχετικά η γραφειοκρατική προσπάθεια η οποία όμω δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Και το άλλο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας ε, των ε, αποδεκτών. Βλέπουμε εδώ μια γλωσσική τροποποίηση. Οι beneficiaries γίνονται recipients. αλλά βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν ε, αυτή την ε, ομοιογένεια που, που χρειαζόμαστε δεν τη βλέπουμε καθόλου. Χαίρομαι πολύ που αφήνεται το θέμα αυτό στις τροπολογίες μας, στον συνάδελφο Ρεβελίνη και εμένα. Επίσης, όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις, σε ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικά θέματα περιμένουμε απαντήσεις στα θέματα αυτά εδώ και χρόνια. Θα ήθελα να σκεφτείτε το εξής, ε, την ε, ε, εξωτερήκευση του ιστορικού κόστους. Βλέπουμε στα τελευταία 5-6 χρόνια ότι η Κομισιόν έχει εγκαταλείψει την ιδέα αυτή πιστεύοντας ότι μπορεί πράγματι να επηρεάσει ε, τις εξελίξεις. Το ότι θέλει να τις επηρεάσει για μένα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ε, θα πρέπει να συνεχιστεί η εξωτερική Ε, τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο ήταν ε, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, η Κομισιόν ε, πιστεύει ότι θα πρέπει να προσέχει να μην χάσει έτσι μεγάλο μέρος του προπολογισμού της. Επίσης, όσον αφορά τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, το πρόβλημα που είχαμε με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το οποίο δεν θα έχουμε στο μέλλον, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποθεί αυτό το θέμα. Ε, υπάρχουν πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα για ε, μας όμως ε, με τη διαδικασία απαλλαγή συνδέεται η υποχρέωση λογοδοσίας της Κομισιόν. Θα πρέπει να εξετάζουμε τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών. Δεν έχει όμως ε, νόημα να έχουμε εκθέσεις 3.000-4.000 ε, σελίδων, ε, οι οποίες όμως να μην έχουν τα στοιχεία που πρέπει να έχουν. Να γνωρίζετε φεύγοντας από εδώ πάντως ότι έχετε την υποστήριξή μας όχι όσον αφορά τις δηλώσεις σας, τις υποσχέσεις σας, αλλά όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσετε. Την τελική απάντηση Κομισιόν και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γκρέσλε συνόψισε πολύ καλά. Το όλο θέμα πρέπει να συνεργαστούμε για τα θέματα που ανάφερα στην ε, εισαγωγή μου. Συμφωνώ απόλυτα ότι η ποιότητα των εθνικών συνόψεων πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Το μελετάμε πολύ το θέμα αυτό και ελπίζω σύντομα να έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Ώστε συμφωνώ ότι η διαφάνεια όσον αφορά τους δικαιούχους πρέπει να διασφαλίζεται. και πρέπει να γίνει, έχουμε περισσότερη εναρμόνιση όσον αφορά τους δικαιούχους. Πολλά έχουμε κάνει, αλλά συμφωνώ ότι το θέμα επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Οι διαπραγματεύσει δεν είναι εύκολες γιατί τρία όργανα παίρνουν μέρος. Πάντως η θέση της Κομισιόν είναι σαφής. Πρέπει να ελέγχουμε τις δαπάνες των κονδυλίων της Ένωσης και από την υπηρεσία αυτή. Κοινό στόχος μας νομίζω είναι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να είναι υπόλογη για το πώς δαπανά τα κοινωτικά κονδύλια. συνοψίζω και εγώ. Είμαι έτοιμος να σας δώσω συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτό που ζητήσατε. Και θα σας πληροφορώ σε τακτική βάση για τις εξελίξεις των πρωτοβουλειών, νέες πρωτοβουλίες. Θα έχουμε στενή συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο Σεμέτα και ας περάσουμε τώρα στο σημείο 5. Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων συστημάτων πληροφορικής σε θέματα ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης. Ο εισηγητής κύριος Μαρινέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να σας παρουσιάσω τις ε, κύριες προτάσεις μου σχετικά με, με τον οργανισμό αυτό. Καταρχήν η δραστηριότητα του οργανισμού. Πολιετής. Χρειάζεται πολιετές πρόγραμμα και χρειάζεται και πρόταση του προπολογισμού πολιετής. και μετά θα προταθούν τα ετήσια προγράμματα εργασίας. Μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλλεται το πρόγραμμα. Το, η Διοικητική Επιτροπή τώρα του οργανισμού. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρότασή μου. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να απαρτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο από 9 μέλη. Δύο να τα προτείνει Κομισιόν, δύο το Κοινοβούλιο και τα πέντε το Συμβούλιο. Και κανένας Ευρωβουλευτής να μην είναι μέλος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Μία απλουστευμένη δομή θα εξασφαλίσει πιο αποδοτική χρήση και μειωμένη δαπάνη, κόστος αυτού του οργανισμού. Επίσης, προτείνω τη σύσταση μιας ελεγκτικής επιτροπής, επιτροπής ελέγχου, τριμελή, τρία μέλη μάλλον από το Διοικητικό Συμβούλιο, που να ασκεί ένα είδος leadership σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Ο οργανισμός θα τον εποπτεύει ο διομεσολαβητής. Δεν υπήρχε πρόταση, γι' αυτό έκανα εγώ μια πρόταση γι' αυτό. Στη μεταβατική περίοδο, μέχρι να οριστεί εκτελεστικός διευθυντής, προτείνω να οριστεί, να διοριστεί μάλλον ένας διευθυντής από την Κομισιόν, υπεύθυνος, ως υπεύθυνος για τον οργανισμό αυτό. Αυτός ο διευθυντής θα είναι αυτός που θα δίνει και τις εγκρίσεις. Αυτές είναι οι βασικές μου προτάσεις για τον οργανισμό. Και αυτό έχει να πει η Επιτροπή μας περί αυτού. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ποιος να θέλει να μιλήσει για την έκθεση του συναδέλφου Μαρινέσκου. Κομισιόν, το Συμβούλιο. Η κυρία Γκρέσλε πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Μαρινέσκο γιατί πραγματικά έκανε κάποιες πολύ καινοτόμες προτάσεις. Για παράδειγμα τη μείωση των μελών στο εποπτικό όργανο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί στους αποκεντρωμένους φορείς έχουμε τελικά περισσότερα μέλη συνήθως. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα νέο δρόμο εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια τέτοια καινοτομία σε κάθε νέο οργανισμό που ιδρύουμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό εδώ να κάνουμε μια δοκιμή και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση γιατί είναι εξαιρετικά καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική δουλειά που έχει κάνει όσον αφορά τις τροπολογίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός των τροπολογιών αυτών είτε αντικατοπτρίζονται ήδη στην παρούσα μορφή του κειμένου αυτού που οριστοκοπήθηκε σήμερα στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, ε, ενώ οι υπόλοιπε. Ε, δεν ε, βλέπω το λόγο η Κομισιόν να μην εξετάσει περαιτέρω θετικά ε, τις τροπολογίες αυτές ε, για το σχέδιο πρότασής της. Ε, οι δύο παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω έχουν να κάνουν με τη σύνθεση του Διαχειριστικού Συμβουλίου καθώς και το θέμα της εσωτερικής ερεκτική λειτουργίας. Έχουμε επιφυλάξεις για τα δύο θέματα αυτά. Καταρχήν όσον αφορά το διαχειριστικό σώμα. Όχι επειδή δεν καταλαβαίνουμε την ανάγκη για αποτελεσματικότητα, επικροτούμε τέτοιες προτάσεις, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή της υπηρεσίας αυτής. θα διαχειρίζεται μεγάλα προγράμματα πληροφορικής, μεγάλα συστήματα πληροφορικής ε, στον, ε, ε, που θα διαχειρίζονται δεδομένα των κρατών μελών, όχι τις υπηρεσίες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ειδικό ενδιαφέρον ελέγχου του τι κάνει η υπηρεσία αυτή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι λογικό κάθε κράτος μέλος να έχει ε, μέλος στο διαχειριστικό συμβούλιο, το οποίο σημαίνει να έχουμε ένα πλήρες διαχειριστικό συμβούλιο ε, όπου να συμμετέχουν όλοι οι χρήστε, διότι αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες ε, των πληροφοριών του συστήματος. Όσον αφορά την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητη η λειτουργία αυτή για να διασφαλίζονται τα συμφέροντα και τα εχέγγυα που θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά την εκτέλεση και τον έλεγχο του προπολογισμού. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η συμμετοχή του, των μελών του Διαχειριστικού Συμβουλίου, των εκπροσωπών δηλαδή των κρατών μελών στην εσωτερική αυτή η ελεγκτική λειτουργία μπορεί να παρεμποδίσουν κάποιες από αυτές τις προσπάθειες ε, που θα πρέπει να είναι αντικείμενο του ε, διαχειριστικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να κλείσω εδώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την πολλή δουλειά που έχει κάνει όσον αφορά τις τροπολογίες. Διότι αυτές αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά που ήδη έχει γίνει. Ε, αντικατοπτρίζουν επίσης τις προθέσεις της Κομισιόν με το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Μαρινέσκου. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Ε, ζητώ συγγνώμη. Όσον αφορά την Διαχειριστική Επιτροπή, εμείς πιστεύουμε ότι το Προεδρείο αυτό θα ε, διαχειρίζεται τα συστήματα ΒΙΣ και Αλλά αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα συστήματα, αυτά τα οποία διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη στη μεταβατική αυτή περίοδο, μέχρι δηλαδή την ε, δημιουργία του οργανισμού. Πιστεύω ότι η Διαχειριστική Επιτροπή δεν ε, θα ασχολείται άμεσα με τη λειτουργία του συστήματος. Το θέμα είναι η εποπτεία που θα γίνεται από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι στη συνθήκη τα κράτη-μέλη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεσπίσει μια τέτοια επιτροπή με τρία μέλη και πιστεύω ότι θα πρέπει έτσι να Μπορούμε να μικρύνουμε το, την ε, Διαχειριστική Επιτροπή αυτής, αυτού του οργανισμού. Όσον αφορά τον ιστορικό έλεγχο, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, αλλά με τις εμπειρίες που έχουμε από άλλους οργανισμούς διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου στην οποία συμμετέχουν κάποια μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορεί, μπορεί να βοηθά τη λειτουργία αυτή και να αποτελεί σύνδεσμο με διάφορες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από εμπειρογνώμονες στον σχετικό τομέα.